για να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο στον κυβερνοχώρο ή τον πόλεμο στο επίπεδο των πληροφοριών. Τονίζουμε επίσης την διαφοροποιούμενη κατάσταση όσον αφορά τους πρωταγωνιστές αυτού του παιχνιδιού, το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης ορισμένων ε, φορέων και μερών, την εμφάνιση δημοφιλών ιστοτόπων που προάγουν την ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας, την διάδοση των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, που είναι και αυτά ιδιαίτερα δημοφιλή. Πολλά λοιπόν έγιναν από τότε στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διάφορους άλλους φορείς αλλά και στην κοινωνία των πολιτών τα τελευταία δύο χρόνια. Στην έκθεση, επίσης, αναφέρουμε αυτές τις δραστηριότητες και τονίζω προκειμένου της, ε, τη σημασία της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, τη σημασία αυτών των πρωτοβουλίων για τη δημοκρατία, καθώς και τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας και της εργασίας με ομοειδάτες χώρες. Στο δεύτερο τμήμα αυτής της έκθεσης διαλαμβανόμεθα των διαφόρων τύπων παραπληροφόρησης και εχθρικής προπαγάνδας και στο τρίτο μέρος Μιλούμε για την προστασία των επικειμένων εκλογών μας, των ευρωπαϊκών εκλογών, των εκλογών του 2019. Το 2019 είναι έτος 29 διαφορετικών εκλογών σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οι ευρωπαϊκές εκλογές βεβαίως που θα γίνουν ταυτόχρονα σε ορισμένες χώρες. Ζήσαμε την προσπάθεια παρίσφρησης της Ρωσική ομοσπονδία σε διάφορες εκλογές και δημοψηφίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και αλλού. Πρέπει λοιπόν να αποδειχθούμε ανθεκτικοί εναντί αυτών των προσπαθειών εμπλοκής. Ο ρόλος της Stratcom East λοιπόν εμπορικημένο θα είναι πολύ σημαντικός και αναφέρουμε και σε δύο άλλες task force. Αναφέρουμε σε αυτήν για τα Δυτικά Βαλκάνια και σε αυτήν για την ε, Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Μίμητσακ μέρος της Αντιπρόεδρου της Κομισιόν, είπα της εκπροσώπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτέ. Σας ευχαριστώ πολύ που διαθέσατε χρόνο για να συζητήσετε ε, αυτά τα ζητήματα παραπληροφόρησης ε, και ξένης παρέμβασης. Πάρα πολύ επίκαιρα θέματα ώψη των ευρωεκλογών. Σας ευχαριστώ όλους ε, για την συνεισφορά σα και ιδίω θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Νίλ Σπιέτα Φωτίγκα που τόσο επίκαιρα κάνει αυτές τις τόσο εύστοχες συστάσεις που συμβαδίζουν με τη λογική και τι δράσεις του σχεδίου δράση κατά της παραπληροφόρηση που υπέβαλε, είπατε, εκπρόσωπος ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ανταπόκρισή μας ε, και η αντίδρασή μας σε αυτές τις κυβερνοαπειλές είναι κοινή δράση. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις προσπάθειές μας, αλλά θα πρέπει και τα κράτη-μέλη συλλογικά να αναβαθμίσουν τις προσπάθειές τους, όπως λέει στα συμπεράσματά του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, στις συστάσεις γίνεται λόγος για το πόσο κομβική σημασία έχει η ελευθερία έκφρασης, ελευθερία λόγου, ο πλουραλισμός ε, για τις ανθεκτικές ε, κοινωνίες διότι οι θεμελιώδεις αξίες μας πραγματικά πρέπει να είναι ε, στο επίκεντρο ε, της μάχης που θα δώσουμε κατά της παραπληροφόρησης. Αυτό είναι ακριβώς το πνεύμα με βάση το οποίο καταρτήσαμε και τώρα εφαρμόζουμε το σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης. Η έκθεση καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξασφαλίσουν ότι η στρατηγική επικοινωνία της Ένωσης θα λάβει ύψιστη προτεραιότητα και ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα συνεργαστούν στενά για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης αυτής. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλα αυτά ήδη συμβαίνουν. Όμως, είναι μια μακρόπνοη προσπάθεια που υπερβαίνει τις ευρωεκλογέ του τρέχοντος έτους. Γι' αυτό και βασιζόμαστε στην συνεχή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από πλευράς δημοσιονομικής. Με το σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης αυξάνουμε τη στελέχωση των τριών ειδικών ομάδων ε, για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, για να μπορούν να ανοιχνεύουν, να αναλύουν και να ε, καταγγέλουν την παραπληροφόρηση, να ευαισθητοποιούν για τον αρνητικό αντίκτυπο, κυρίως όμως ε, να βελτιώνουν τον τρόπο επικοινωνίας και μετάδοσης των αξιών και των πολιτικών μας. Την επόμενη εβδομάδα θα δρομολογηθεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, όπως λέει το σχέδιο δράσης, ένα σύστημα που θα καταστήσει πιο εύκολο για τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν εκτιμήσεις, δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης εν ώψη των ευρωεκλογών. Αυτό θα βελτιώσει ε, την ευαισθητοποίηση θα προωθήσει κοινέ δράσει, κοινή αντίδραση εφόσον χρειαστεί, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αύξηση τη ευαισθητοποίηση και την μεγαλύτερη ανθεκτικότητα τη κοινωνία. Εκτιμώ το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το έργο ε, των ειδικών ομάδων Stratcom και σε ό,τι αφορά ε, την επικοινωνιακή πολιτική και τη μάχη τους κατά της ε, παραπληροφόρησης. Για τα Δυτικά Βαλκάνια ε, και το Νότο επίσης έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά αυτές οι ειδικέ ομάδες. Η Stratcom έχει καταλογοποιήσει, έχει αυξήσει να για πάνω από 5.000 περιπτώσεις παραπληροφόρησης από ρωσικές πηγές. Δυστυχώς αυτός ο αριθμός ε, θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα πολύ περισσότερο. Δεν θα ε, φύγει το πρόβλημα αυτό, δεν θα λυθεί σύντομα από ό,τι φαίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουν απαλλαγμένε από ξένε παρεμβάσει οι ευρωεκλογέ και ένα τρόπο να το πετύχουμε αυτό είναι ε, αυξάνοντα την ευαισθητοποίηση για τι προκλήσει ε, που υπάρχουν με στενή συνεργασία με τα μίντια, κοινωνία των πολιτών, πλατφόρμε μέσων κοινωνική δικτύωση μεταξύ άλλων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση εργάζεται σε πλήρη συντονισμό με το Κοινοβούλιο και τι υπηρεσίε της Κομισιόν. Φυσικά, το σχέδιο δράση θα σεβαστεί πλήρω τι εθνικές προσεγγίσει, την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία ε, των μέσων ενημέρωση που θα καθοδηγούν τι δράσει μα. Ταυτόχρονα, βελτιώνουμε τη συνεργασία μα για την αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων και υβριδικών απειλών με τους διεθνού μα εταίρους, όπω είναι το ΝΑΤΟ και η ομάδα των 7, το G7 συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Ήδη εξελίσσεται. Ανταλλάσσουμε εκθέσεις εκτίμησης ε, για το περιβάλλον των πληροφοριών. Ε, συντονισμένες δράσεις αναλαμβάνουμε. Ασκήσεις ε, με σενάρια κάποιων ευρυδικών απειλών. Επίσης, θα πρέπει να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο με τι γείτονε χώρε για να προωθήσουμε το θεματολόγιο τη Ένωση. Θέλουμε να επενδύσουμε στη θετική επικοινωνία, στη δημόσια διπλωματία στις χώρες γειτονία. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση και να προωθήσουμε τις κοινέ αξίες και τα κοινά συμφέροντα. Η δημόσια διπλωματία και η στενή συνεργασία με τις αποστολές αντιπροσωπής της Ένωσης ε, επιτόπου είναι πολύ ισχυρά εργαλεία που προβάλλουν μια θετική εικόνα της Ένωσης στον κόσμο. Το καλύτερο αντίδοτο στην παραπληροφόρηση αφενός είναι ένα υγιές περιβάλλον ε, για τα μέσα ενημέρωσης και αφετέρου η προβολή των ε, θετικών ενωσιακών πολιτικών. Οι πολίτες μας έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση σωστές πληροφορίες, όχι ψευδείς ειδήσει. Έχουν το δικαίωμα σε ένα πλουραλιστικό δημοσιογραφικό περιβάλλον, σε ποιοτικέ πληροφορίες. Γιατί μιλάμε για την ποιότητα της δημοκρατίας μας, για την ποιότητα της Ένωσης μας. Ευχαριστώ. E, e, Ευχαριστούμε Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστούμε την κυρία Φωτέγκα για την ε, εξαιρετική της έκθεση. Είναι ένα κείμενο που αναγνωρίζει την ε, σημασία των εξτρατιών προπαγάνδας και της ανάγκες να τις καταπολεμήσουμε. Ιδίω όπου υπάρχει κατασκοπία από τρίτες χώρες. Πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφορία μεταξύ των 100 ε, μελών και προσπάθειες σωστής ενημέρωσης. Ο πόλεμο στο επίπεδο τη πληροφόρηση είναι ε, περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Πρέπει να δράσουμε γέρο και να μην ξεχνάμε ότι. Ο Καζίμοφ μίλησε ήδη από το 2013 για την ε, σημασία και το πόσο επίκαιρο είναι το ψηφιακό επίπεδο στην ό,τι αφορά τα πολεμικά πράγματα. Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να διαχωρίζουμε σωστά τα ψεύδια από την αλήθεια. Γιατί είναι ένα νέο τρόπο να διεξάγεται πόλεμο. Και μάλιστα έλεγε ο ίδιο ότι υπάρχουν κάποιοι που χρησιμοποιούν όλο το ταλέντο σε αυτό το επίπεδο για να πετύχουν του πολεμικού του σκοπού. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε συνεννόηση και με το ΝΑΤΟ και το G7 για όλα αυτά τα θέματα. Το να παραμείνουμε αδρανείς θα σημαίνει απειλή εις βάρος 500 εκατομμυρίων πολιτών και υπονόμευση των αξιών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε και τώρα ε, ε, τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ο κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο παραπάνω από δύο μήνες ε, γίνονται εκλογέ στην Ευρώπη και όπως και με το Brexit, με την εκλογή του Αμερικανικού, Αμερικανού Προέδρου ή την εκλογή του Γάλλου Προέδρου, ε, υπάρχουν προκλήσεις και σε αυτή την περίπτωση και σίγουρα στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, υπάρχει το πρόβλημα της παραπληροφόρησης, ε, προπαγάνδας και των ψευδών αυτών ειδήσεων που θα κατακλείσουν, που θα μεταφέρουν πληροφορίες προπαγάνδας και θα είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε ξεχωρίσει κανείς το ψέμα από την αλήθεια ε, την πληροφορία από την ε, προπαγάνδα και νομίζω ότι πραγματικά είναι σημαντικό που ασχολείται με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων η ΕΕΔ. Αυτό όμως είναι ένα πρώτο βήμα. Το πρόβλημα εγώ που βλέπω είναι ότι η τεχνολογική ε, πρόοδος μας έχει ξεπεράσει κατά πολύ όπως και συνεχίζει να κάνει. Ε, εμείς ε, προσπαθούμε να παλέψουμε με προχθεσινά μέσα και όπλα τη χθεσινή παραπληροφόρηση, ενώ η προπαγάνδα έχει προχωρήσει πιο πέρα. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τι είναι ήδη στην αγορά και πώς θα είναι το μέλλον και υπάρχουν ε, δυσκολίες κανείς ε, να διακρίνει ένα βίντεο αν είναι ε, κατασκευασμένο, αν είναι πραγματικό ε, και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση θέλω να ευχαριστήσω όλους τους και όλους που συνεργάστηκαν για την εκπονησή της. Είναι τελευταία φορά που βρίσκομαι εγώ εκπρόσωπος της Αυστρίας χάρηκα πολύ αυτά τα πέντε χρόνια ε, και θα ήθελα ε, να μην ε, επηρεαστεί και να μην φρεναριστεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση από εθνικιστικές ή αντιευρωπαϊστικές τάσεις. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εκ μέρους της ΕΣΥΑΡ, κύριος Τσαρνέσκι. Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, συγχαρητήρια στην κυρία Φορτάκα για την εξαιρετική έκθεση. Εμείς είμαστε οι μπροστοφυλακοί, ξέρετε, όσον αφορά το θέμα. Και όταν είσαι μπροστά, έτσι είναι τα πράγματα. Έχεις έναν χώρο, ο οποίος είναι επιδεκτικός εκμετάλλευσης από όσους δίνουν τη μάχη κατά της ελευθερίας υποκινούμενοι πολλές φορές από τρίτες χώρες που δεν αξίζει καν να αναφέρω. Στην πολιτική ζωή έχουμε όμως ευκαιρία να κάνουμε κάτι. Έχουμε εκλογές. Και το Brexit μπορεί να είναι μια ευκαιρία για αλλαγή. υπάρχουν και άλλες συγκυρίες οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για μας. Ξέρουμε βέβαια ότι υπάρχουν ευκαιρίες και για τους άλλους. Ευκαιρίες που θα αξιοποιήσουν, θα εκμεταλλευτούν οι εχθροί της ελευθερίας, οι εχθροί της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα, εκ μέρου των φιλελευθέρων, ο κύριο Αυστριβίτσιος. Πρόεδρε, κύριε Πιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόσβαση στην πληροφορία είναι όλο και πιο επικίνδυνη, πιο επιδεκτική σε ψευδοειδήσεις. Τα κρατημέλικοι κυβερνήσεις συνεχίζουν να αγνοούν ή να αρνούνται την ύπαρξη εχθρική προπαγάνδα. Πρέπει επιτέλου να γνωρίσουμε το πρόβλημα, να αξιολογήσουμε την απειλή στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβουμε μέτρα με τρόπο δραστικό για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι ψευδοειδήσει. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τα ψέματα, την προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση, τις ψευδοειδήσεις, όλα αυτά που προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διαφόρων ειδών τρομοκρατίες. Υπάρχει στρατιωτική τρομοκρατία, υπάρχει τρομοκρατία κατά της κοινωνικής συνοχής. Λοιπόν, Όλα αυτά είναι απειλέ κατά τη δημόσια τάξη. είναι απειλέ κατά των αξιών και τη ζωής των δικών μας κοινωνιών. Και όλα αυτά συνδέονται με τον υβριδικό πόλεμο κατά των κοινωνιών μας, κατά της καρδιάς και του μυαλού των πολιτών μας. Δίνουμε λοιπόν μια μάχη. Έχουμε μια μάχη μεταξύ εξωτικών, μεταξύ ψευδοειδήσεων, αόρατων εχθρών και το πρώτο βήμα που κάναμε ήταν η Stratcom, η Stratcom για να αντιμετωπίσουμε τις ψευδοειδήσεις. Χρειάζεται να λάβουμε αποφάσεις γρήγορα μέσω αυτής της ομάδας Cruise, ε, η οποία πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με ακόμη περισσότερα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα για τους πράσινους η κυρία Ρεμπέκα Χάνος. Κύριε αξιότιμε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, οι εκπρόσωποι των ομάδων στις διαπραγματεύσεις ε, της ε, Έκθεση ε, της δεύτερης χέρα ήταν ε, πολύ πιο ε, σύμφωνη σε σχέση μεταξύ του σε σχέση με την επεξεργασία της πρώτης έκθεσης. Τώρα θέλουμε να καταπολεμήσουμε την προπαγάνδα και τη ρητορική μίσους και στις ε, περισσότερες ε, περιπτώσεις ε, η χώρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η Ρωσία που έχει θύμα όχι μόνο την Ουκρανία αλλά το Κρεμλίνο κάνει όλο και περισσότερες προσπάθειες με όλο και περισσότερα μέσα να επηρεάσει τους Ευρωπαίους πολίτες κατά των κυβερνήσεών τους με τελευταίο παράδειγμα τις διαμαρτυρίες των κίτρινων γυλαίκων κατά των μεταναστών. Υπάρχει λοιπόν παρότρινση ε, και επίσης ε, επηρεασμό της κοινή γνώμης ε, και για το Brexit μεταξύ άλλων. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε γιατί κατά την άποψή μου θα πρέπει να οργανωθεί πολύ περισσότερο η πληροφόρηση, η σωστή πληροφόρηση, να δοθούν περισσότερα χρήματα και οι υπηρεσίε των κρατών μελών και οι σχετικές αρχές να συνεργάζονται και και με το ΝΑΤΟ και με τις μυστικές υπηρεσίε, αλλά ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζονται ανεξάρτητα μίντια. Ο πλουραλισμός στις δημοκρατικές κοινωνίες είναι το α και το ω κατά του μίσους, ε, κατά της προπαγάνδας. Ε, επομένως, εδώ πρέπει να δώσουμε τη βάση μας. Ευχαριστώ. Kaso για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια από την ε, υποβολή αυτής της έκθεσης. Ε, δεν φαίνεται γιατί έχουμε τα ίδια επιχειρήματα, τις ίδιες καταγγελίες ε, που έχουν ξεγυμνωθεί εδώ και δεκαετίες, σχέσεις, καλής κοινωνίας, και τα λοιπά και βλέπουμε ότι υπάρχει η ίδια βούληση τα λάθη των ιστορικών πολιτικών να τα ρίχνουμε σε ξένους παράγοντες. Ενώ το εκλογικό σώμα είναι αυτό το οποίο τιμωρεί τα πλειοψηφικά κόμματα για τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους και το αποκορύφουμε ότι περιλαμβάνεται στο Ισλαμικό κράτος μια αναφορά που το μόνο που κάνει είναι να χειροτερεύει τις σχέσεις μας με την Ρωσία. Ε, γιατί τη συγκρίνει ουσιαστικά με μια τρομοκρατική ομάδα που καταδικάζει ο ΙΕ. Μιλάμε για δίωξη των δημοσιογράφων. Ε. Μιλάμε για ανεξάρτητη δημοσιογραφία που χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα είναι ανεξάρτητη. Βλέπουμε ότι η Ένωση ε, ασκεί μόνο κριτική, αλλά δεν ασκεί καμία κριτική σε αυτά που ίδια κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Καστάλτο, ευχαριστώ. Συνάδελφοι, είναι αναντήρητο ότι οι υβριδικές απειλές, κυρίως στον τομέα της πληροφόρησης, αποκτούν στρατηγική σημασία για τις κοινωνίες μας. Ιδίως τώρα που τα νέα τεχνολογικά μέσα έχουν αναπτύξει την ε, ταχύτητα και την ένταση των επιθέσεων σε διεθνές επίπεδο με την ε, ε, αλληλοδιασύνδεση που προκύπτει. Όμως, συνάδελφοι, θα πρέπει να κοιτάξουμε, να προστατεύσουμε από τις ψευδείς ειδήσει τους πολίτες, αλλά να μην τους αφήσουμε εκτεθειμένους σε τρίτους ε, τρομοκράτες ή κράτη ε, στην όλη προσπάθεια μας. Θα, θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και την παραπληροφόρηση αλλά και τις απειλές του τζιχάντο ε, online με τον ίδιο τρόπο, με τους κανόνες μας. Θα πρέπει στον τομέα αυτό να μην παραμείνουμε στα τόσα λίγα που έχουν γίνει, ιδίω από τα κράτη που χρησιμοποιούν μέσα πολέμου, πρόξη όπως λέγονται. Θα πρέπει λοιπόν να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στη γεωγραφική διάσταση, γιατί κάποιες φορές είναι ασαφής η ορολογία που χρησιμοποιείται και μερικές φορές μάλιστα είναι και στα όρια της ε, λογοκρισίας. Θα πρέπει λοιπόν να επιβάλλονται κυρώσεις ε, αμερόληπτες και αποτελεσματικές. Ιδάλλως δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σοφοζέρ για την ε, Ευρώπη των Εθνών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Φωτίγκα, δεν ασχολείστε με τη στρατηγική επικοινωνία στην πραγματικότητα. Προτείνετε μέτρα κατασταλτικά για να καταπολεμήσετε μια σαφή προπαγάνδα η οποία προέρχεται από δίθεν εχθρικέ χώρε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σα εμπνέει, η ίδια λογική τη συνωμοσιολογία και των Μπολσεβίκων, τη απειλή των Μπολσεβίκων, όπω τη κυρία Καλνιέτε. Εδώ οποιαδήποτε αντίρρηση στο φιλευρωπαϊκό Εχείρημα εγχείρημα το βλέπετε ως προπαγάνδα. Ε, ε, τα κίτρινα γυλαίκα είναι ε, πίσω του η Μόσχα. Το Brexit το Πούτιν. Βρέχει στην Βαρσοβία φταίει ο Πούτιν. Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε με το κεμαλαϊκισμό που κατακλείζει την Ευρώπη. Φαίνεται να έχετε σταλινιστικές αιμονές. Πότε θα ξαναρθούν τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Εδώ λέτε ότι είναι προδότε όσοι δεν συμφωνούν με αυτέ τι ιδέε. Προδοσία είναι να ε, θέλουμε να εργαστούμε για μια Ευρώπη χριστιανική που θα συνεργαστεί και με τη Ρωσία για να τη δημιουργήσει. Που θα εμπνέεται για έναν κόσμο ο οποίο θα λειτουργεί ε, χωρίς καμία ψυχή. Τι θέλετε, η Ευρώπη να μην έχει ψυχή ούτε ρωσική ούτε καμία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος... Έχετε λάβει γαλάζια κάρτα. Από τον κύριο Τάραντ. Τη δέχεστε. Κύριε Τάραντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σοφοζέρ, συμφωνείτε μαζί μου ότι το να συγκρίνετε την κυρία Καρνιέτε με το σταλινισμό και όλα τα άλλα που είπατε είναι κάπως ε, μη αρμόζων διότι όπως εγώ γνωρίζω γεννήθηκε σε σιβηρικό γκούλαγκ. Είναι μια πλήρωτη, απαντήστε. Παρακαλώ. Ε, κοιτάξτε, ε, χθε ε, συζήτησα με την κυρία Καλνιέτε και γνωρίζω για τις εμπειρίες της από το Κούλακ. Δυστυχώς δεν με άκουγε ενώ μιλούσα. Και τη είπα ότι ως προς τη Ρωσία θα πρέπει να παρέμβουμε όχι μόνο λόγω συγκινησιακών ε, καταλήπων ή από ε, εκδικητικότητα, αλλά αναλύοντας ψυχρά και αντικειμενικά την κατάσταση. Και μπορώ να πω ότι και εγώ πολέμησα κατά του κομμουνισμού και ότι το 89 εδώ στο Στρασβούργο συγκεντρώσαμε όλες τις αντικομμουνιστικές δυνάμεις πριν την πτώση του τείχους. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Σοφοζέρ αλλά πρέπει να συνεχίσουμε την ε, διεξαγωγή της συζήτησής μας κανονικά. Ο λόγος στον κύριο Φουντούλη για ένα λεπτό. Ας πούμε μια φορά την αλήθεια μέσα σε αυτή την αίθουσα. Δεν σας ενοχλεί η προπαγάνδα, κύριε της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άλλωστε, από την ίδια την Ένωση εκπορεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό προπαγάνδας που κατευθύνεται προς τους πολίτες. Σας ενοχλεί μόνο οτιδήποτε στρέφεται εναντίον των δικών σας συμφερόντων η ένωση χρηματοδοτεί εκατοντάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες προπαγανδίζουν τα ιδεολογήματα των κρατούντων αυτή τη στιγμή σχηματισμών. μάλιστα είχατε το θράσος να βαφτίσετε τις δικές σας πεποιθήσεις ως αξίες της ενώσεως χωρίς ποτέ βέβαια να ερωτηθούν οι πολίτες των κρατών μελών για κάτι τέτοιο. το χειρότερο όμως είναι πως με τη στάση σας αυτή αποδεικνύεται το γεγονός πως θεωρείτε τους πολίτες ανίκανους να κρίνουν τις πληροφορίες που δέχονται και να επιλέξουν τις θέσεις που τους εκπροσωπούν αντίθετα με μια πατερναλιστική λογική θεωρείτε πως μόνο εσείς μπορείτε να τους υποδείξετε τη σωστή εντός εισαγωγικών άποψη. για εσάς οι πολίτες είναι ελεύθεροι να ψηφίζουν ό,τι θέλουν αρκεί να συμφωνεί με εσάς. για εμάς οι πολίτες της ένωσης έχουν το νου και τη γνώση να κρίνουν και να αποφασίζουν ποιος τους αντιπροσωπεύει. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν υπάρχει μία σύσταση που θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά, θα ήταν κατεπηγόντως η ομάδα δράσης για τα θέματα της Ανατολικής Γειτονίας να γίνει μια διαρκής, ε, ένα όργανο που να λειτουργεί διαρκώς με την απαραίτητη χρηματοδότηση και το απαραίτητο προσωπικό, την απαραίτητη επάνδρωση στελέχωση. Θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Ευρωπαϊ... την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για τη Δημοκρατία, ε, το καταπίστευμα δηλαδή, για να υπάρξουν ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ε, και ε, αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό. Θα πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίση να είναι ε, διαφανεί ω προ τι δωρεέ που δέχονται. Θα πρέπει να ξέρουμε ποια κόμματα απευθεία ή εμέσω ε, ε, χρηματοδοτούνται από τι ρωσικέ μυστικέ υπηρεσίε ή τι μεγάλε εταιρείε τη Ρωσία, του μεγάλου ομίλου, για να γίνουν τα παραθυράκια από που θα μπορούν να προωθήσουν τα όχι και τόσο δημοκρατικά του συμφέροντα εκείνοι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η κυρία Γουόρντ για ένα λεπτό. Η προπαγάνδα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλώς για ακροδεξιούς ευρωσκεπτικιστές που έχουν ε, γεννηθεί και μεγάλα τραφεί εδώ και θέλουν να καταστρέψουν το όνειρο ειρήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανακάλυψε όταν εργάστηκε για την έκθεση του 2016 για το θέμα αυτό, έχει να κάνει με τη Ρωσία και τις χώρες που δεν συμμεριστούν στις ευρωπαϊκές αξίες αυτό το θέμα. Ε, επηρεάστηκε το ε, ψήφισμα το 2016 από τις υπηρεσίες του Πούτιν και αυτές του οι δράσει μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο και στι επερχόμενε ευρωεκλογέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να λάβει μέτρα αυστηρά. Θα πρέπει να ε, ε, υπάρξουν περισσότερα εργαλεία από τι τεχνολογικέ εταιρείε για τον εμπλουτισμό τη προπαγάνδα και να γνωρίζουμε κατά την ταυτότητα όσων χρησιμοποιούν τι πλατφόρμε. Να σβήνονται τα σχόλια που ε, δεν ξέρουμε τι οικονομικά συμφέροντα τα στηρίζουν. Επίση, χρειαζόμαστε περισσότερη ευαισθητοποίηση σε πολιτικό επίπεδο. Λόγω χάρη, ο κύριο Γάλλο ακροδεξιό βουλευτή, έκανε δώρα στην κόρη του Πούτιν και στον εκπροσωπό του εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτά θα πρέπει να απαγορεύονται. Επίση, ε, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αγνοεί την εχθρική προπαγάνδα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια τη προεκλογική εξετρία για τον Brexit. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε τα ε, χρήματα από την παραοικονομία και όλα αυτά που χρηματοδότησαν αυτήν την εκστρατεία. Σα ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να παραμένετε στο χρόνο μιλία σα και τώρα για ένα λεπτό ο κύριο ε, Κρίστιαν Πρέντα. Ευχαριστώ. Η αντιμετώπιση της προπαγάνδας ε, προαπαιτεί το να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς της προπαγάνδας. Και διαφέρουν αυτοί από τη μια χώρα στην άλλη. Στη Ρουμανία, λόγου χάρη, ένας πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός διαδίδει ψεύδι υποστηριζόμενος από έναν αξιωματικό του κοκκινού στρατού, πρώην αξιωματικό του κοκκινού στρατού. η κυβέρνηση λοιπόν να διαδίδει ψεύδι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο ο μηχανισμός επαλήθευσης των ε, ειδήσεων που χρέωσε το Υπουργείο να πάρει θέση και να πει ε, εντάξει πρόκειται για ε, νοθευμένες ειδήσει τελικά. Ε, κακικό έλεγχο των ε, πηγών. Η κυρία Νταντσίλε, επίση πρωθυπουργό, είναι στη Σπούτνικ κάθε εβδομάδα. Πολλοί πολιτικοί έχουν καταδικαστεί για διαφθορά και υπάρχει. γίνεται κουβέντα για το πώς απειλεί το κράτος δικαίου της χώρας ο Τζόρτ Σόρος και πώς επίσης είναι κακό πράγμα η δημοκρατία στη Ρουμανία. Αυτό αρχίζει να κατακλείσει την κοινή γνώμη. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο κάθε χώρα όπως και στη δική μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ο μιλητής ο κ. Πιτσούλα για να λεπτό. Ε, Cambridge Analytica, Το σκάνδαλο της Cambridge Analytica απλώς επιβεβαιώνει πως ε, μπορούν να επηρεαστούν εκλογές και δημοψηφίσματα. Αναμένουμε βεβαίως περισσότερη ενημέρωση από το Λονδίνο να δούμε πραγματικά ε, τι συνέβη και με τον Brexit. Δεν μπορούμε λοιπόν να υποτιμήσουμε την εμπλοκή της παρεμβάσεις των Ρώσων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμούμε την απειλή. Ίσα ίσα πρέπει να δούμε τι γίνεται στα Βαλκάνια, τι γίνεται με τις υποψήφιες χώρες. Φυσικά δεν είναι μόνο η Ρωσία. Οι ψευδοειδήσει προέρχονται και από δυτικέ πηγές αλλά και από αλλού. Ο στόχος τους όμως είναι ένας, να καταλύσουν τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε τώρα λίγο πριν από τις εκλογές να δώσουμε αληθή πληροφορία στου πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το υπαριθμό 1. Ευχαριστώ. Κύριε Σκόβατσεφ. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Σκόβατσεφ, Αντιμετωπίζουμε όντω υβριδικό πόλεμο. Πρέπει να λάβουμε μέτρα. Τα εφιστάμενα μέτρα δεν είναι επαρκή. Η East Stratcom η ομάδα κρούσης, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, να γίνει μια ανεξάρτητη ενισχυμένη διεύθυνση με επαρκή χρηματοδότηση. Στη Βουλγαρία έχουμε μια τέτοια υπηρεσία υπό την Μαρία Γκάμπριελ. Η βουλιαρκή κυβέρνηση πρότεινε τη δημιουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας η οποία θα ενισχύει την ερευνητική δημοκρατία και η οποία θα πατάσει την παραπληροφόρηση και η οποία γενικότερα θα ενισχύει όλους τους φορείς που διεξάγουν πόλεμο κατά των ψευδοειδήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μείνει στο απειρόβλητο πρέπει να καταλάβει πού υστερεί σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε. Κύριος Γκάλερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στον συνόλεφο Άγγεν Φρόιντ. Συμφωνώ απόλυτα με το 100% των όσων είπε. Αυτό θα του έλεγαν ήταν εδώ, δεν είναι εδώ. Βέβαια, δεν κατάφερε μέσα σε δύο λεπτά να πει ούτε μια φορά τη λέξη Ρουσία. Ρωσία. Δεν ξέρω, ίσω να είναι αυστριακή ιδιαιτερότητα. Τέλο πάντων, τα πράγματα όμω πρέπει να τα λέμε με το όνομά του. Ε, η Ρωσία το μόνο που θέλει να καταφέρει είναι η αποσταθεροποίηση τη Ευρώπη. Ε, να αποδυναμώσει το mainstream. Όλα τα άλλα είναι ελκυστικά. Οι Τικεή που η, η τότε ΣΣΕΔΟΥ η τώρα Ρωσία είχε τη δική της ειδολογία έχουν περάσει. Και η ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας πρέπει να ενισχυθεί. Εκεί που πέφτει το χρήμα, ε, κύριε ε, Σαφάζερ, ε, πρέπει να υπάρξουν νόμοι για να μην επιτρέπεται η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα. Μπορεί να παίξει ένα συντονιστικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η ομάδα ειδική είστε στρατκόμ πρέπει να ενισχυθεί και να υπάρχουν και οι απαραίτητες επαφές και διαδικασίες δικτύωση με εθνικούς συνδέσμους από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Ρανζέλ που είναι ο εμόδιο επόμενο ομιλητή. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον επόμενο, τον κύριο Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σοβαρή απειλή στη κατά τη Δημοκρατία. Πώ θα αντιδράσουμε αποτελεσματικά κατά της προπαγάνδας, παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων από τρίτε χώρε, Όλο και πιο δύσκολα μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό Πρέπει λοιπόν και σε εθνικό και σε νοσιακό επίπεδο να προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε τις αξίες μας και να αντιμετωπίσουμε τον κυβερνοπόλεμο και τον υβριδικό πόλεμο. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι ε, όμορες χώρες προς Ανατολάς και προς Δυσμάς και προς Νότον. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε στο περιφερειακό επίπεδο, να βελτιώσουμε την επικοινωνία πάνω στα θέματα που απτούνται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητώ επίσης ε, μεγαλύτερη χρηματοδότηση, περισσότερη στελέχωση, περισσότερα μέσα ε, και περισσότερη συνεργασία ε, με τις επίσημους χώρες όπως είναι η αντιπροσωπή της Ένωσης στις τρίτες χώρες. Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, της εχθρικής προπαγάνδας πρέπει να είναι προτεραιότητα, όχι μόνο για τις ευρωεκλογέ αλλά και ε, εν ώψη και το ε, επερχόμενου Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν. Πρέπει καλύτερα να μεταδώσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αλλιώς οι δημοκρατίες μας μπορεί να μην ανθέξουν, να μην επιβιώσουν απέναντι στις εξωτερικές αυτές απειλές και πιέσεις. Ευχαριστώ. Κύριος Κέλαμ είναι επόμενος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, το Stratcom έχει δώσει καταπληκτικά αποτελέσματα ε, με 5.000 παραδείγματα να λέει στατιστικά το τι συμβαίνει. Αυτή η ομάδα δράσης λοιπόν του Stratcom θα πρέπει να γίνει μόνιμη ομάδα με τις δικές της, με δικά της κονδύλια και το δικό της προσωπικό. Εδώ λοιπόν ε, θα πρέπει να ε, δώσουμε το πλήρες νόημά του στο Στράτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σημαντική αρμοδιότητα για να βελτιώσει τις δεξιότητες και να δώσει τη δυνατότητα απόκρισης ε, στα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία με τον ιδιωτικό κλάδο, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη και να προωθήσουμε την εκπαίδευση κατά της παραπληροφόρησης. Θα πρέπει να δώσουμε κατά απαραίτητα κονδύλια στο Stratcom. Θα πρέπει να αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συντονίσει τις σχετικές προσπάθειες με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Στέτινα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Εδώ έχουμε 38 συστάσεις την έκθεση. Ο στόχος όμως όλων είναι να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα κρατών. Στο 8, στο προήμιο επίσης, αναφέρονται κύριες πηγές ε, παραπληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2014 ο Ρώσος στρατηγός Σίμωφ θέσπισε νέες μορφές πολέμου στον κυβερνοχώρο λέγοντας ότι αν επιλέξουμε σωστά τις λέξεις και τις διαδώσουμε με το σωστό τρόπο, ο πόλεμος αυτός θα έχει πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα από τις βόμβες και τις ρουκέτες. Λοιπόν, ας ξυπνήσουμε επιτέλους και ας συνειδητοποιήσουμε ότι χάνουμε τον κυβερνοπόλεμο με τη Ρωσία. Ας πούμε επιτέλους τη, τα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αλλιώς θα χάσουμε σύντομα τις δυνατότητές μας σε αυτόν τον χώρο. Ευχαριστώ. Ε, δεν βλέπω. Ε, κυρία Αντρικένε. Όχι, δεν είναι εδώ. Σουίτσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με απασχολεί το θέμα των ψευτοειδήσεων και της παραπληροφόρησης. Ακούμε τόσο πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία. Κυρίω για τον ρόλο τρίτων χωρών. Λοιπόν, εγώ ανησυχώ και πρέπει όλοι να ανησυχούμε για την κατάσταση. Γι' αυτό είμαι υπέρ τη έκθεσης. Θα υπερψηφίσω γιατί διαλαμβάνεται των δυνατοτήτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση και τι ψευδοειδήσει. Μπορούμε να κάνουμε πολλά σε εθνικό επίπεδο, όμω το διαδίκτυο είναι παγκόσμιο. εννοείται ότι συμβαίνει, συμβαίνει παντού, πέραν των σύνορων. Η προπαγάνδα από την Ανατολή είναι επίφοβη, σίγουρα επηρέασε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στον Εμένο Βασίλειο, τα αποτελέσματα του οποίου φυστάμεθα σήμερα. Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι Βρετανοί πολίτες. Ό,τι και να λέμε. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να πατάξουμε την προπαγάνδα από τρίτους φορείς, από τρίτες ε, χώρες, ιδιαίτερα εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών. Ευχαριστώ. Ζροεύσκη. Πρόεδρε. Στην αρχή της θητείας μας είχα πει δύο λόγια για τον ευρυδικό πόλεμο. Είχα πει ότι ευρυδικός πόλεμος σημαίνει ευρυδική εμπλοκή, ευρυδικά μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση, αλλά να διασφαλίσουμε και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη σωστή εκπαίδευση και την απαραίτητη συνεργασία. Στρατηγική συνεργασία θα έλεγα. Δυστυχώ είμαι σήμερα απογοητευμένο από τα όσα έχει κάνει, μάλλον δεν έχει κάνει η Κομισιόν, διότι ήδη το 2016 είχαμε ζητήσει από την Κομισιόν να κάνει περισσότερα κ. Φορτέγκα είχε αναλάβει πρωτοβουλίες στην Επιτροπή Άμυνας. Η Κομισιόν θα πρέπει να είναι μπροστά από τους διάφορους παίκτες στον χώρο, στον πόλεμο της παραπληροφόρησης, του πολέμου στον κυβερνοχώρο. Δυστυχώς η Κομισιόν τώρα τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και μάλιστα αποκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση σε προβλήματα τα οποία ήταν γνωστά στο δημόσιο χώρο εδώ και χρόνια. Οι περίπου 40 συστάσεις είναι καλές εν πάση περιπτώσει, είναι επίκαιρες. Ας κάνουμε κάτι τώρα, χωρίς καμία καθυστέρηση παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Προσέλκυση προσοχής του Προέδρου. Έχετε το λόγο κύριε Ρανζέλ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που άργησα κύριε Πρόεδρε, αλλά ε, είχα μια συνάντηση με τον κύριο Μπαρνιέ. Καταλαβαίνετε ότι ήταν σημαντικό αυτό και δεν μπορούσα να είμαι εδώ βέβαια. Θα ήθελα κυρίως να πω το εξή. Το θέμα της προπαγάνδας, όλος ιδιαίτερος της προπαγάνδας που στόχο έχει να εξαπατήσει την κοινή γνώμη και όπως γνωρίζουμε συμβαδίζει με την όλη, πάει εν παραλίλω με τις συζήτηση που κάναμε για τις ψευδεί ειδήσει. έρχεται από συγκεκριμένε χώρες. Και εδώ πρέπει να έχουμε μια πολύ αποφασιστική ε, δράση. Να αναχαιτήσουμε κάθε προσπάθεια, τα στρατηγικά συμφέροντα, τα οποία συνήθως είναι κακοπροαίρετα από τρίτες χώρες να επιβληθούν και να επηρεάσουν τις δικές μας προεκλογικές εκστρατείες, τις συζητήσεις μας και το υποψηφίσματά μας. Γι' αυτό λοιπόν η ε, στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή η καταπολέμηση αυτού του είδους των προσπαθειών, είναι πολύ σωστή. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ευρυδικός πόλεμος δεν είναι κάτι το καινούριο. Ωστόσο, οι εξελίξεις έχουν επιταχυνθεί. Έχουν ε, ανοίξει νέοι διαβλοί και ακόμα περισσότερο μέρος του κοινού μπορεί να πέσει θύμα προπαγάνδας, γιατί υπάρχει πρόσβαση πιο εύκολη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι προσπαθούν να, να επηρεάσουν τις δημόσιες συζητήσεις στην Ευρώπη, τη δημοκρατία, ε, γιατί έχουν περισσότερο χρόνο για να... χώρο για μάλλον για να δράσουν. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω ότι στηρίζω θερμά τι συστάσει αυτή τη έκθεση. Και παρόλο που σε μια ανεπτυγμένη δημοκρατία θα πρέπει να είναι σαφέ, δεν είναι. Ε, θα πρέπει να υπάρχει και επικριτική ε, δυνατότητα κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, η κριτική μπορεί να είναι και επικοδομητική, δεν είναι κάθε κριτική ε, εχθροπραξία. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ και πολύ καιρό δεν ακούμε τι φωνέ των πολιτών. Θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσει που να εξυπηρετούν και τα δικά του συμφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Επιτίδιο. Ε, στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την αλματώδη εξέλιξη τη τεχνολογία, οι αρχέ και οι μέθοδοι τη προπαγάνδα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν με πολλού και διαφόρου τρόπου, οι κυριότεροι από του οποίου είναι η παραποίηση τη αλήθεια και η διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ε, βασική αρχή για μια δημοκρατική κοινωνία να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ε, εχθρική προπαγάνδα είναι η παρουσίαση της αλήθειας στο κοινό και όχι η δίωξη των πολιτικών αντιπάλων και των δημοσιογράφων οι οποίοι ασκούν ε, κριτική στην κυβέρνηση η παρουσιάζουν διάφορα σκάνδαλα. σε εθνικό επίπεδο η ενημέρωση του κοινού η αντικειμενική και αμερόληπτη επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ενός λειτουργικού συστήματος ραδιοτηλεοράσεως πολλές φορές όμως το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί σωστά. αυτό συμβαίνει στην ελλάδα που η ραδιοτηλεόραση εθνική έχει μεταβληθεί σε όργανο κομματικό του κυβερνώντος κόμματος και μάλιστα φτάνει στο σημείο να μην καλεί στις εκπομπές τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές του κόμματος στο οποίο ανήκω της χρυσής αυγής που είναι η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. όπως αντιλαμβάνεσαι με τέτοιες μεθόδους υπάρχει αναξιοπιστία και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε εχθρική προπαγάνδα. ευχαριστώ. E, Ευχαριστούμε. Ροχόνεν Λέρνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα κοινωνικά μέσα και στα παραδοσιακά μέσα η παραπληροφόρηση είναι εξίσου ε, απειλή κατά της δημοκρατίας. Γι' αυτό οι πληροφορίες και οι ειδήσει που λαμβάνουμε πρέπει να είναι ακριβείς και αληθεί. για να μπορούν και οι άνθρωποι να αποφασίζουν σωστά όταν πρόκειται να ψηφίσουν ε, με περιστατωμένη γνώση και επίγνωση. Θα πρέπει λοιπόν όταν εντοπίζονται οι ψευδεί ειδήσει και παραπληροφόρηση στα κοινωνικά δίκτυα, να απαιτείται και να απομακρυνθούν, να σβηστούν. Θα πρέπει να εντοπίζονται ω δυνατόν γρηγορότερα προτού ε, διαδοθούν ε, ευρέως. Θα πρέπει οι πλατφόρμες στο διαδίκτυο να, να καταστήσουν σαφές ότι και οι κανόνες της διαφήμισης που, τη στηρί, που του στηρίζει θα πρέπει να είναι διαφανείς θα πρέπει να μην μπορούν να μετακινούνται τεράστια ποσά μεσολογαριασμών ε, τόσο γρήγορα και τα τεχνολογικά μέσα αλλάζουν διαρκώς. Είναι πολύ εύκολο να στήσει κανείς ένα ψεύτικο βίντεο και ένα ψεύτικο φιλμάκι και οι ψευδείς ειδήσει πρέπει να καταπολεμηθούν με την ε, σωστή ε, γνώση, με τον αλφαβητισμό των μέσων μας και ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Μαριάς κύριε πρόεδρε συζητούμε εδώ για την παραπληροφόρηση την προπαγάνδα τις ψευδείς ειδήσει αλλά αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και εναντίον του ίδιου του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου διότι όπως ξέρετε όλοι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ανέθεσε σε μια δημοσκοπική εταιρεία να κάνει δημοσκόπηση για τις ευρωεκλογέ η οποία δημοσκοπική εταιρεία αντί να κάνει δημοσκόπηση πήρε τις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο δημοσκοπήσεις που έγιναν για εθνικές εκλογές και έβγαλε συμπεράσματα για το ποιοι εκλέγονται και ποιοι δεν εκλέγονται από αυτή εδώ την ευρωβουλή πόσοι ευρωβουλευτές από εμά δεν θα εκλεγούν και πόσοι δήθεν θα εκλεγούν. αυτό είναι μαύρη προπαγάνδα παραμονές των ευρωεκλογών είναι fake news είναι καθοδηγημένη προπαγάνδα εναντίον συγκεκριμένων ευρωβουλευτών. αυτό πρέπει να καταγγελθεί και να απαγορευτεί και να σταματήσει αυτή την τακτική το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διότι είναι έσχος και γι' αυτό πρέπει να τοποθετηθείτε όλοι συνάδελφοι να μην επιτρέπουμε τα fake news ότι ορισμένοι δίθεν από εμά δεν θα εκλεγούν επειδή το λέει μια δημοσκοπική εταιρεία και αυτό έχει αναπαραχθεί σε όλα τα μίντια σε όλη την ευρώπη. είναι ντροπή είναι έσχος. Ευχαριστώ πολύ για το παθιασμένο αυτό σας λόγο και τελευταίο στο Catch the Eye, Κάρσκι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολλοί είπαν για την παραπληροφόρηση μέσω παραδοσιακών και νέων μέσων ενημέρωσης παραπληροφόρηση έχουμε και εδώ, στο Ευρωκοινοβούλιο, στο πλαίσιο της συζήτηση. Ένας από τους δράστες είναι ο κύριος Σαφοζέρ, που βρώμησε ε, το στόμα του χρησιμοποιώντας ε, ε, το, βάζοντας στο στόμα του το όνομα του Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου ντροπή και όνειδος και είπε ότι δεν τηρούνταν οι συστάσεις ε, και τα όσα είπε και τα κηρύγματα του ε, Ιωάννη Πάρτου δεύτερο. Αυτό πραγματικά είναι ανήθικο. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς που λένε αυτά. Και φαντάζομαι θα του τα μεταφέρουν το κύριο Σαφοζέρ αυτά που λέω. Μπορεί να μείνει ε, αυτή η ομιλία ε, ως μία από τις ε, πιο εντυπωσιακές, αλλά είναι αποτέλεσμα, είναι προπαγάνδα και παραπληροφόρηση ουσιαστικά. Να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Νίμιτσα για να ολοκληρωθεί έτσι η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Εξαιτήμα βουλευτέ. Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Φωτίγκα και του βουλευτέ ε, για τι παρεμβάσει του. Από αυτή τη συζήτηση, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχουμε ένα κοινό ε, συμφέρον και ενδιαφέρον να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της ε, ξένης παρέμβασης και της παραπληροφόρησης ε, ενώπιον των ε, ευρωεκλογών. Είναι λοιπόν αυτή η συζήτηση και μια ευκαιρία για να προβάλλουμε περισσότερο το θέμα και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση. Ολοκληρώνοντας, θέλω να επαναλάβω για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες μου για τον ρόλο του Κοινοβουλίου που έχει βάλει προτεραιότητα το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Φωτίγκα, για να κλείσουμε. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Εδώ μιλούμε για τον δηλητηριασμό των ψυχών των πολιτών μας. Το καλύτερο παράδειγμα ήταν η κατηγορία της χαρά της ε, και μου της ιδέας. Πούτιν ο ίδιος συνεχίζει τις πολιτικές του Στάλιν και το λέει. Το λέει ο ίδιος χωρίς περιστροφές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους κοιόδης εισηγητές για τις συνεισφορές τους. Όλες εξαιρετικές. Είχαμε ουσιαστικό διάλογο για το θέμα σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα, χάρη στη δική σας συνεισφορά, θα βοηθήσει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν την εχθρική προπαγάνδα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ, ο οποίος με βοήθησε σε πολύ δύσκολες στιγμές όταν εγώ αντιμετώπισα μεταξύ άλλων και κάποια προβλήματα υγείας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Εδώ κλείνει η συζήτηση επί του θέματος, η ψηφορία αύριο. Και τώρα, επόμενο θέμα, επόμενο σημείο στη μίληση διάταξη και είναι η συζήτηση για το Αφγανιστάν. Σύσταση της κυρίας Φωτιγκά και πάλι για τη Συμφωνία συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη. Έχουμε εδώ μία έκθεση τη κύρια Φωτίγκα για τη Συμφωνία συνεργασία, όπως προείπα, μεταξύ ευρωπαϊκή Ένωση και Αφγανιστάν. Δίνω τον λόγο στην εισηγητήρια την κυρία Φωτίγκα. Παρακαλώ, δίνω τον λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Επιτροπέ, κυρίε και κύριοι, Η Συμφωνία Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη υπεγράφει τον Φεβρουάριο του 2017. Εν μέρη, θα έλεγα, και προσωρινά τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου του 2017. Το Συμβούλιο αποφάσισε να παραμείνει μεικτή συμφωνία, δηλαδή να εμπλακούν και τα κρατημέλη στην κύρωση της συμφωνίας. Η κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν παραμένει δύσκολη. Και όμως, μόνο το 56% της επικράτειας παραμένει υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων, το οποίο σημαίνει ότι μόνο το 65% του πληθυσμού απολάβει της κυβερνητικής προστασίας. Το 2002 ξεκίνησε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτοτε πάνω από 3,66 δισεκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστικής βοήθειας χορηγήθηκαν στη χώρα ακολούθησε μια δεκαετία προσαρμογής, αλλαγών, μέχρι λίγο πολύ το 2014 και σκοπεύουμε να ξέψουμε άλλα 1,4 δισεκατομμύρια για να σταθεροποιήσουμε το Αφγανιστάν. Σε συνδυασμό με την νατοική δύναμη ΙΣΑΦ. Και χάρη στην υποστήριξη και άλλων χωρών συμπεριλαμβανομένης της δικής μου. Όλοι μαζί εργαστήκαμε για την ασφάλεια στην περιοχή αν και με την εμφάνιση του ISK, του ΤΕΣ, του, του ISIS δηλαδή μετά από τα γεγονότα στο Ιράκ. Η εμφάνιση λοιπόν αυτών των δυνάμεων στην περιοχή αποσταθεροποιούν την περιοχή στο έπακρο. Η κοινή πολιτική εστιάζεται στο κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου, την σταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών, τη σταθεροποίηση υγεία της περιοχής, την σταθεροποίηση της κοινωνίας, προκειμένου θέλω να συγχαρώ όλους τους συμπλεκομένους για τόσα επετεύχθησαν στην περιοχή. Και όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στις θεριστικέ. Η πρόσβαση, ας πούμε, στις υπηρεσίε υγείας χάρη στην ευρωπαϊκή βοήθεια από το 9% Πήγαμε στο 57%. Μια τεράστια βελτίωση το προσδόκιμο ζωής από τα 45 έτη ανέβηκε στα 60 έτη. Η εκπαίδευση επίσης. Η συμμετοχή στις εκλογές. Η συμμετοχή των γυναικών. Όλα αυτά βελτιώθηκαν όλα αυτά κάτι σημαίνουν για τη χώρα. Η συμφωνία υπεγράφει από την Φιτρικά Μογκερίνη, την υπατή εκπρόσωπο και την πρόεδρο τη Επιτροπή και τον Υπουργό Οικονομικών του Αφγανιστάν, παρουσία του Πρόεδρου της χώρας. Εμείς ως βουλευτές λυπούμεθα πραγματικά, διότι οι σχετικέ λεπτομέρειε όσον αφορά τη διαπραγμάτευση τη συμφωνία έφτασαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη καθυστέρηση. Μετά, ουσιαστικά εκ των υστέρων, μετά την υπογραφή τη συμφωνία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλέψει τη συνθήκη όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, είμαι υπέρ συμφωνία, υποστηρίζω, υπερψηφίζω και ελπίζω ότι θα υπερψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε και τώρα εκ μέρου της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο λόγος στον Επίτροπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε και κύριοι, επιτρέψτε μου